της Συνόδου τον Ιούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 78 μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου υπέγραψα οκτώ νομοθετικά κείμενα σύμφωνα με την κανονική νομοθετική διαδικασία έχουν εγκριθεί. Τους τίτλους λοιπόν μπορείτε να τους βρείτε στα πρακτικά της συνεδρίασης αυτής. Και τώρα κυρίες και κύριοι σας παρακαλώ να λάβετε